Περάμε τώρα σε ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Θα ήταν οι πιο σύντονες συνδόσεις αυτή τη στιγμή, γιατί <laughs> μισή ώρα ξεπέρασαμε το συνεδρίες και πρέπει να τελειώσουμε 8.30 για να μπορέσουν οι ειρηνείς να ξεπροστούν και να συνεχίσουν στις 9. Λοιπόν, χωρίς περαιτέρω εισαγωγή, Περνάμε στην ενότητα υπαριθμού 17. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη κι εγώ. Το έγγραφο στο οποίο αναφέρθηκε ο εξάτιμο ε, κύριο Βουλευτή δεν είναι ένα έγγραφο που έχει υιοθετηθεί από την Επιτροπή και δεν έχει εγκριθεί η δημοσίευσή του. Πρόκειται για ένα έγγραφο που εξολογεί το κόστος και τα ωφέλη της μείωσης κατά 30% των εκπομπών. Ήταν μια πρόταση, μια ανακοίνωση που πρότεινε το Συμβούλιο Περιβάλλοντος 17 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Δεν πει μόνο και το χρόνο για να προεδρεθούμε. Πρόκειται όμως για μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση για την γνώμη μας. Και κατόπιν θα υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες που θα πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερώς. Εκτός αυτού η ανεκκίνηση αυτή υπευλήθηκε μέσα στα πλαίσια της οδηγίας ETS, μια ανάλυση δηλαδή της κατάστασης των τομέων που είναι ε, ευαίσθητοι για τη χρήση της ενέργειας και σύμφωνα με τα κριτήρια της Κομμενχάης Θα ήθελα να σας πω πολύ σαφώς ότι δεν είναι η πρόθεση της Κομισιόν να πάρουμε μια απόφαση την επομένη μετά την παρουσίαση της ανακοίνωσης αυτής να περάσουμε στα 30% πρόκειται για ένα βήμα για να φροντίσουμε ότι όταν κάνουμε τη συζήτηση για τη μείωση αυτή, τότε θα μπορούμε να έχουμε καλά ενημερωμένη βάση για να προχωρήσουμε από εκεί στις συζητήσεις μας. Αυτός είναι ο στόχος των ερωτήσεων. Ανάλυση, στοιχεία, κόστος, υπολογισμούς για να έχουμε πραγματικά ενημερωμένη συζήτηση και θα ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσει και θα συμμετάσχει και το κοινοβουλίο στη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Τσίρκο. 30 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αναφέρεται στο εγγράφο αυτό ότι όταν ε, πρόκειται να επιτευχθεί αυτός ο νέος στόχος θα υπάρχουν και επιδράσεις στην ε, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή λέει ότι κάποιοι χρηματοδοτικοί πόροι θα χρειαστούν που θα προέθουν από τα διευθυντικά ταμεία των κρατών. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα υπάρχει μια απλή μεταφορά κονδυλίων Παραδείγματο χάρη όσον αφορά την υποδομή και τι οδικέ μεταφορέ, Εκεί, από εκεί θα αφαιρεθούν ίσω και οι πόροι. Η έχει το λόγο. Ευχα... Ελπίζω ότι ο κύριος βουλευτής θα σεβαστεί το γεγονό ότι δεν μπορώ να πάω στι λεπτομέρειε αυτή, γιατί αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία αναφέρεται στην ανακοινωσία, δεν ήταν σωστό. Και κατά τη διάρκεια τη ακρόασή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα πει ότι εμείς θα πρέπει να λέμε ότι όταν χρησιμοποιούμε χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φροντίζουμε τα διάφορα σχέδια, αναφερθήκατε στην υποδομή, να ελεγχθούν ανάλογα με το κατά πόσο είναι συμβατά με την προστασία του κλίματος. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό και αν θα καταφέρουμε έτσι να κάνουμε και μείωση 30% μέχρι το 2020. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ανάλυση και να καλέσουμε μεταξύ άλλων τους βουλευτές και το Συμβούλιο να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Πρώτα σε ευχαριστώ. Έχω δύο σημαντικές ε, ερωτήσεις. Η κυρία Τίκαου και ο κύριος Δέβης. Πρώτη κυρία Τίκαου. Τρία λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εμείς ψηφίσαμε μια έκθεση σήμερα για την ε, τροποποίηση της οδηγίας που αφορά την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας σε κτίρια. Αυτή είναι μια απαρχή μια νέας διαδικασίας ε, στα πλαίσια της θα μπορούσαμε να μειώσουμε την ε, κατανάλωση της ενέργειας και τις εκπομπές εξ αυτού στα κτίρια. Και χρειαζόμαστε γι' αυτό όμως χρηματοδότηση και ελπίζω να υπάρχει αύξηση των ποσοστώσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέιβις. Πρόεδρε, επιτρέπε. Η αρχική πρόταση δεν αντιμετωπίζει την κλίμακα του θέματος που αντιμετωπίζεται. Πολλοί από του βουλευτέ εδώ και πολλέ από τι κυβερνήσει του Βουλή δεν αποδεχόνται την ανάγκη κατεπηγόντων μέτρων για να αποφύγουμε την κλαματολογικέ αλλαγή. Είναι πολύ εύκολο να υπογράφει κανένα εφολογικά ψηφίσματα. Τώρα όμως που πρέπει να περάσουμε σε πρακτικές λύσεις, δεν θα πρέπει εσείς να αντιμετωπίσετε το θέμα διαφορετικά και άμεσα. Καταρχήν θα ήθελα να μελετήσω αυτή την ε, πρόταση που γίνεται σήμερα για την ενδεικτική απόδοση των κτηρίων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει κάτι αυτό. Υπάρχουν και κάποια νέα μέσα που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όντως ώστε εκείνοι που ε, ασχολούνται με τα κτίρια να μπορούν να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας. Ε, ε, θα το εξετάσω ευχαρίστω γιατί συμφωνώ με την ερωτήση σα ότι ένα από του τομεί όπου πολλά μπορούμε να κάνουμε τα κτίρια είναι ακριβώ μέσα στα πλαίσια τη αποτελεσματική χρήση ενέργεια και κυρίως όσον αφορά την απόδοση των κτηρίων. Είναι πολύ τεράστιο θεματικό και είναι πραγματικά γελίο ότι χρησιμοποιούμε και σπαταλούμε ενέργεια που δεν ωφελεί κανέναν. Όσον αφορά τον Κριστέρης έχω να πω Το εξή. Εγώ προσπάθησα να δω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όταν φτάσουμε εκεί. Γιατί παρόλε στι συζητήσει, ιδίω στο ΕΒ που είχαν μια τεράστια συζήτηση του θέματος, εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα πρέπει ίσως να διορθώνονται κάστοτε τα προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει τίποτα που να είναι αντίθετο με τα κύρια αποτελέσματα της επιστήμης. Ότι πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το θέμα, πρέπει να είμαστε σοβαροί όσον αφορά αυτό και υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους και οι σκεπτικιστές του κλίματος θα πρέπει να συμφωνήσουν με εμά και θα πρέπει να κάνουμε κάτι με, για την ενεργειακή απο, απόδοση. Και αν δεν προχωρήσει η Ευρώπη εδώ φοβούμαι ότι θα χάσουμε, θα χάσουμε πολύ τις αναψώμενες αγορές αυτού του αιώνα στους ανταγωνιστές μας. Οι διαρροές άνθρακα δεν είναι τόσο προβληματικές γιατί αν κάνουμε πράγματα που θα οδηγήσουν στην απώλεια θέσεων απασχόλησης, πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί ακριβώς όταν διστάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και χαίρομαι που βλέπω ότι φαίνεται η νέα Βρετανική κυβέρνηση είναι πολύ φιλόδοξη όσον αφορά το θέμα αυτό των κλιματολογικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Πρώτα σε ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση, υπαριθμό 18 της κυρίας Γκέργη του Όντεμπεργκ για τις δράσεις επιτροπής των δομέων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα ήθελα καταρχήν να στραβώ στον Επίτροπο Πανιέ για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκέρνικα Τουίτεμπερκ για την ερώτησή σας που βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το διαδίκτυο. Ε, καμιά φορά τα δικαιώματα αυτά της της ε, ιδιοκτησίας ε, θεωρούν ότι είναι ένα εμπόδιο για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς. Δεν είναι σωστό αυτό γιατί αυτό επιτρέπει ε, στους ε, ε καλλιτέχνες ε, να πουλήσουν αν θέλετε το προϊόν τους και αυτό ισχύει και όχι μόνο για τους καλλιτέχνες αλλά και για την βιομηχανία κλπ και με το απόδοση μπορεί να συνεχίσουν οι άνθρωποι αυτοί να δημιουργούν και άλλα έργα. Αυτό είναι ένα πρότυπο που υπάρχει εδώ και εκατοντάδες ετών. Βέβαια η διαχείριση των δικαιωμάτων έχει εξελιχθεί λόγω της εξέλιξης των τεχνηλιών που έχουν φτάσει σήμερα από το ραδιόφωνο και τηλεόραση στην, στο διαδίκτυο. Κάθε φορά που υπάρχουν νέα οικονομικά μοντέλα αλλάζει η μορφή της εκμετάλλευσης ε, των δικαιωμάτων αυτών και τους πράσπισης επίσης των δικαιωμάτων. Εγώ αυτό που θέλω να προστατεύσω είναι να, τη δημιουργία, προσπαθώντας να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέα οικονομικά μοντέλα. Στις 13 Ιανουαρίου το είπα αυτό στην ακρόαση ενώπιον ημών και αυτό που θα κάνω είναι ακριβώς να εξετάσω μαζί σας ε, το θέμα αυτό. Η ψηφιακή ατζέντα που υιοθέτηκε στις 19 Μαΐου η Κομισιόν πέρσι ήταν πάρα πολύ σημαντική και σήμερα θα έχω τρία μέτρα. Δηλαδή, καταρχήν μια πρόταση οδηγία για την συλλογική διαχείριση των ανθρωπικών δικαιωμάτων που θα επιτρέψει στις ενότητες αυτές να οργανωθούν καλύτερα για να μπορούν να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στο διαδίκτυο και μονοθετική διαχείριση Επίσης, ε, όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων διακυβέρνησης, διαφάνειας, για να επιστραπεί έτσι η δημιουργία, ο καθορισμός μιας τιμής και να υπάρχει μια απόδοση πιο διαφανής. Δεύτερον, μια οδηγία για τα ορφανά έργα που δημιουργεί την απαραίτητη νομική ε, προστασία για την ε, ψηφιακή μετατροπή σε βασικούς ε, φορείς των ε, έργων της ε, Ευρωπαϊκής Παράδοσης. Τρίτον, θα πρέπει να, ο, να λύσουμε τους όρους δημιουργίας νέων υπηρεσιών, βίντεο και λοιπά στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε θα εμπλακούμε σε όλα τα θένα που προβλέπουν μια διαχείριση προστινέμενης αξίας στο διαδίκτυο για να δούμε πώς διακρινίσουμε τους ε, κανόνες, να δούμε ποιο λόγο παίζει η τεχνολογία για την ε, αναγνώριση και την απόδοση των έργων αυτών και πώς θα μπορούμε να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί και να καταπολεμήσουμε ιδιαίτερα την, την πειρατεία στο διαδίκτυο και την μαύρη οικοδομία εμείς θέλουμε μια Ευρώπη που επιτρέπει τη δημιουργία νέων οικονομικών μοντέλων. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα πρέπει να γίνει. Νομοθετική παρέμβαση ή άλλη. Παρ' αυτά δεν έχω καμία αυταπάτη όσον αφορά στην ανάγκη να βρούμε λύσεις. Δεν θα υπάρχει μια λύση για όλους, αλλά θα είναι καλό να ξαναδημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά και να έχουμε μια πραγματική οικονομική πολιτική για τον πολιτιστικό τομέα της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Η κυρία Οντεβέκ, μια συμπληρωματική ερώτηση. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, Πολλέ πρωτοβουλίε έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για την πράσινη βίβλο του 2008, για τα συγγραφικά δικαιώματα, για τα δικαιώματα των δημιουργών. Έχουμε ένα προαιρετικό σύστημα εξαιρέσεων. Και δεν λειτουργεί, δεν διευκολύνει την κατάσταση. δεν υπάρχει και μάλιστα ευνοεί την, ε, όσους αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα και όχι τους πραγματικούς δημιουργούς. Ε, θα πρέπει να υπάρξει σημείο ισορροπίας. Έχουμε διάφορες εξαιρέσεις και για τις βιβλιοθήκες και για όσους έχουν προβλήματα όρασης και ούτω καθεξής. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Επιτροπή για αυτό το θέμα των εξαιρέσεων ως προς το δικαίωμα των δημιουργών. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να σας επιβεβαιώσω ε, κάποια πράγματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν επιλέξαμε να λειτουργήσουμε βάσει του άρθρου 118 της συνθήκης θέλουμε να έχουμε μια άδεια πανευρωπαϊκή για την προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού. Θεωρούμε ότι έτσι θα είναι πιο αποτελεσματική η προστασία της δημιουργίας. Η πράσινη βίβλος αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και θα πρέπει πράγματι να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά τα θέματα, όπως για παράδειγμα είναι οι εξαιρέσει για όσους έχουν προβλήματα όρασης. Για να είναι αποτελεσματικός αυτός ο τίτλος του Ευρωπαίου δημιουργού, αν θέλετε, του Ευρωπαϊκού Δικαιώματος Προστασίας της Δημιουργίας, θα πρέπει πρώτα να εκχωρηθεί από από την εθνική κυριαρχία και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το δεχθούν τα κράτη-μέλη από πλευράς πολιτισμικής, εθνικής, νομικής ή και άλλης. Και άλλωστε και να γινόταν δεκτό κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να ισχύσει για ε, έργα παλαιότερα, αλλά για έργα π.χ. μουσικά τα οποία θα συντεθούν στο μέλλον, από εδώ και στο εξής. πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένη διατύπωση βεβαίως και για τα ορφανά έργα, αυτά τα οποία αποκαλούμε ορφανά έργα, θα, σας, θα διαβουλευτώ μαζί σας και θα ζητήσω τη γνώμη όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Ίκο. Ε, ε, Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον προβλέπετε την αναθεώρηση της οδηγίας για το copyright στην κοινωνία της πληροφορία. Και το λέω αυτό διότι χρειαζόμαστε μια νομική ασφάλεια. Ε, δυστυχώς οι εξαιρέσεις ερμηνεύονται διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν διαφορετικές αποφάσεις ε, στα κράτη-μέλη και για το λόγο αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας κάτω από το πρίσμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. <coughs> Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Προς το παρόν δεν έχουμε πρόθεση να τροποποιήσουμε τον κατάλογο των εξαιρέσεων έτσι όπως προβλέπεται στην οδηγία του Bilbao. Νομίζω ότι έχουμε υιοθετήσει μια προοδευτική, ρεαλιστική προσέγγιση με τις τρεις πρωτοβουλίες για τη ε, ορφαλά έργα για την πράσινη βίβλο και για τη συλλογική διαχείριση. Αυτές είναι οι τρεις προσεγγίσεις μας. Τις εξήγησα. Δεν θα τροποποιήσουμε τον κατάλογο με τις εξαιρέσεις. Δεν είναι στις προθέσεις μας προς το παρόν. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στο ερώτηση επαριθμό 19 για, του Άλαν Κέλλη για τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Καλωσορίζω την κυρία Μάλμστρομ, η οποία θα απαντήσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μου ζήτησε ο κύριος Αλμούνια να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Δεν βλέπω τον κύριο Κέλλη. Α, μπορείτε να μου τον δείξετε. Α, εκεί είστε. Με ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη για την ερώτηση που μας απευθύνεται. Για να υπάρξει συνέχιση στην ε, περιφερειακή ανάπτυξη ε, αποφασίστηκε να ισχύσουν τα προβλεπόμενα για όλη την περίοδο 2007-2013 ε, για την ανάπτυξη των περιφερειών και τις ε, ε, κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, αναγνώρισε η Επιτροπή ότι θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές όπου αυτό είναι απαραίτητο. επομένω, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να δίδεται στα κράτη-μέλη να κάνουν ενδιάμεση αναθεώρηση του χάρτη ενισχύσεων αναλόγως με τις περιφέρειες βάσει του άρθρου 137 εδάφιο Γ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρία από τα 17 κράτη-μέλη που ήταν ενδιαφερόμενα επαφάσισαν τελικά να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι και το ίμιση των περιφερειών που είναι επιλέξιμε με νέες περιφερειές τις οποίες θα ορίσουν εκ των υστέρων. Οι συνθήκε συνθήκες μπορεί να αυξηθεί και η ενίσχυση των περιφερειών που ήδη έχουν οριστεί ω επιλέξιμε βάσει του ε, χάρτη πορεία. Η επιλεξιμότητα των νεοριστησών περιφερειών αλλά και η αύξηση των ενισχύσεων αξιολογούνται με βάση το μέσο όρο έτσι όπως έχει φανεί στα πρόσφατα ε, στοιχεία της Eurostat για τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα ποσοστά απασχόλησης και ούτω καθεξής. Επομένως στόχος είναι οι κρατικές ενισχύσεις να στοχεύουν προς την οικονομική ανάπτυξη των μειονεκτούντων εθνικών περιφερειών, μειονεκτούντων σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της ίδιας χώρας. Οι τρεις αυτές χώρες ε, αποφάσισαν να γνωστοποιήσουν τις τροποποιήσεις που έχουν κάνει σε αυτό το χάρτη και δείχνει όλο αυτό το πράγμα ότι ε, η οικονομική κρίση δεν έχει πλήξει τόσο σημαντικά ε, τις περιφέρειες αυτές. Ευχαριστώ, κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Το βρίσκω εντυπωσιακό ότι μόνο τρία κράτη-μέλη έχουν ε, κάνει αίτηση και αυτό είναι απίστευτο. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή όπου χάσαμε χιλιάδες ε, θέσεων εργασίας ε, και 3.000 περίπου και σήμερα 800 θέσεις εργασίας χάθηκαν από την Pfizer. 300 στην περιοχή μου που είναι στο νότο της Ιρλανδίας. Μιλάμε για το ότι η κατάσταση ελπίζω να αλλάξει, γιατί αν δεν αλλάξει αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει ενεργά μέτρα έτσι ώστε να προσελκύσει μεγάλες εταιρείε. Αυτό είναι αρνητικό και πρέπει να αλλάξει. Περιμένω λοιπόν από την Κομισιόν να ακολουθήσει διαφορετική στρατηγική γιατί εγώ πιστεύω ότι ο χάρτης κρατικών ισχύσεων είναι απαρχαιωμένος. Επίτροπος. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, όπως είπατε και εσείς, ίσως να είναι περίεργο το ότι μόνο τρία κρατημέλη ζήτησαν αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αυτή όμως είναι η κατάσταση, όπως δείχνουν τα στοιχεία σήμερα το πρωί. Πολλά κρατημέλη και πολλές ε, περιοχές ε, πλήττονται από την οικονομική κρίση. Ίσως όμως ορισμένα κρατημέλη να θεωρούν ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Γιατί όπως είδαμε, πολύ λίγα μέλη ζήτησαν κάτι τέτοιο η δυνατότητα προσφέρθηκε σε 17 κρατημέλη, αλλά μόνο τρία ε, δραστηριοποιήθηκαν. Και φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι ο κύριος στόχος του μακροχρόνου προγράμματος είναι να έχουμε συνέχεια για τις ε, περιοχές ε, και υπάρχουν βέβαια και άλλα μέσα για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Όμως είμαι σίγουρη ότι η Επίτροπος κύριος Αλμούνια θα συζητήσει το θέμα μαζί σας αργότερα. Επόμενη ερώτηση του 20 του κύριου Πόσελτ ε, σχετικά με την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ουκρανίας σε επίπεδο αστυνομικών αρχών. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ για την ερώτησή σου για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η συνεργασία αυτή, η συνεργασία διασυνοριακή, ε, αυτό καταρχήν είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη διμερή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ουκρανία, κυρίως μέσα από τη λειτουργία της Europol. Στις 4 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους ε, υπήρξε μια συμφωνία ε, με την Europol και την Ουκρανία και αυτή επιτρέπει το συντονισμό των εργασιών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Η στρατηγική συμφωνία δεν επιτρέπει την ανταλλαγή ε, προσωπικών στοιχείων για υπόπτους. Αυτή μπορεί να λάβει χώρα μόνο με χώρες ε, που έχουν λειτουργική συμφωνία με την Europol. Και πριν ολοκληρωθεί μια τέτοια συμφωνία, η Ουκρανία ε, πρέπει να επικυρώσει τη συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορά στην ε, προστασία των ε, ατόμων και των δεδομένων. Αυτά όλα εμπίπτουν στις προτεραιότητες Κομισιόν που επιθυμεί η Ουκρανία να έχει προστασία των δεδομένων με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτό θα επιτρέψει να υπάρχει ε, μια ανεξάρτητη αρχή ε, η οποία και θα στηρίζεται ε, τεχνικά και με εμπειρογνωμοσύνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ε, τη συνεργασία με την Ουκρανία και μέσα από αποστολές στήριξης Πέρυσι η UBAM σε συνεργασία με τη Frontex, την OLAF και άλλες πρωτοβουλίες στήριξαν τις ε, συνοριακές, τους συνοριακούς ελέγχους ε, ε, συνεργασία και με τη Μολδαβία για να αντιμετωπιστεί το έγκλημα στα σύνορα και η λάθρομετανάστευση. Ο κύριος Πόσελτ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την πολύ καλή απάντηση. Ήθελα μόνο να ρωτήσω τι θα γίνει τελικά με την υποστήριξη της εκπαίδευσης των αστυνομικών. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ε, ανατολικής ε, της συνεργασίας προς Ανατολάς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ε, Αστυνομική Ακαδημία συμμετέχουν ή αυτό γίνεται μόνο σε επίπεδο κρατών μελών. Κοιτάξτε, με την Ουκρανία έχουμε ένα μόνιμο διάλογο για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Στέφαν Φιούλε, ο συνάδελφός μου, έχει παρουσιάσει ε, το πρόγραμμα της συνεργασίας, συμμετέχω βέβαια και εγώ, ε, καλύπτονται εσωτερικά θέματα για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις Ουκρανικές αρχές να προχωρήσουν ε, σε αυτά τα θέματα για πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας. Και αυτό θα εξεταστεί σε μία συνάντηση με τις Ουκρανικές αρχές μετά από λίγες εβδομάδες. Η συνεργασία δεν προβλέπεται για το άμεσο μέλλον. Αυτό όμως μπορεί να συζητηθεί από τη στιγμή που η Ουκρανία έχει προβεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί τους, είναι ένας σημαντικός ε, γείτονας ε, και γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλό για μας αν θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε περαιτέρω. Βεβαίως και οι Ουκρανοί πρέπει να βελτιωθούν, εμείς όμως είμαστε πρόθυμοι να τους ε, βοηθήσουμε για να δούμε τι τελικά θα γίνει μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στην ερώτηση παριθμών 21 του κυρίου Παπα-Νικολάου για την έκρηξη της εγκληματικότητας στην Ευρώπη. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Μαραθώνιος για μένα. Πρέπει να απαντήσω σε πολλές ερωτήσεις. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Ευρωστάτ δημοσιεύτηκαν στις 29 ε, Μαΐου της περασμένης χρονιάς και καλύπτουν την περίοδο μέχρι και το 2007 και δεν φαίνεται εκεί καμία έκρηξη της εγκληματικότητας. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι βεβαίως και υπάρχει θέμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να ε, προλάβει και να εφαρμόσει τα δέοντα ώστε να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα στην Ευρώπη. Αυτός ο στόχος είναι μέρος του προγράμματος δράσης της Στοκχόλμης για την οικοδόμηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη. Ένα πρόγραμμα δράσης που θα υλοποιηθεί τα επόμενα ε, πέντε χρόνια. Νομίζω ότι προλίγου η συνάδελφος κυρία Ρέντιν ήταν εδώ και συζήτησε μαζί σας, σας ανέλησε διεξοδικά το πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης. Από εκεί και πέρα και πέρα από αυτά θα έχουμε μια ανακοίνωση για την ε, στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια και θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιολόγηση των απειλών για τα επόμενα πέντε χρόνια και θα ε, συμπεριληφθεί σε αυτή τη στρατηγική ε, το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιούν αποτελεσματικά όλα αυτά τα εργαλεία οι, όλες οι αρχές δημόσιες και ιδιωτικές. Έχουμε το εμπόριο ανθρωπίνων όντων, το κυβερνό έγκλημα και την κλοπή των ταυτοτήτων. Αυτά είναι πράγματα που αφορούν όλες τις χώρες και γι' αυτό εμείς ως Επιτροπή θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και σε νομοθετικό επίπεδο. Και θα το κάνουμε αυτό συνεργαζόμενοι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Πρέπει να ε, συντονίσουμε ε, δράσεις, διάλογο, ε, κατάρτιση, έρευνα για να αυξήσουμε την αμοιβαία αναγνώριση. Συνεργασία με τρίτες χώρες. Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία αυτή για να καταπολεμήσουμε σωστά και αποτελεσματικά την εγκληματικότητα. Ε, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι ε, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για να είμαστε φιλόδοξοι θα πρέπει να υπάρχει βούληση πολιτική από πλευράς κρατών μελών. Και όλα αυτά εξαρτώνται και από τους εθνικούς πόρους που αφιερώνονται για την επίτευξη των στόχων. Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει με χρηματοδοτικά προγράμματα τα κράτη-μέλη ώστε να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και άλλωστε η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει και πολλές αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για τα θέματα αυτά. Έχετε και εσείς ευθύνη, έχετε σημαντικό ρόλο ε, για την οικοδόμηση ενός χώρου ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ε, πέρσι είχαμε μια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είχα συμμετάσχει στη σύνταξη της έκθεσης αυτής και είχα ε, υπογραμμίσει τη σημαντική αύξηση των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ και των 200 ευρώ. Δηλαδή χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο αυτά τα χαρτονομισμάτα για νομιμοποίηση παράνομων προσόδων και εσόδων. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτσι ώστε να φανεί να διερευνηθεί ποιος τελικά χρησιμοποιεί αυτές τις πολύ μεγάλες ποσότητες των ε, χαρτομισμάτων των 500 ευρώ. Ίσως χρησιμοποιούνται για φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή ή διάφορες άλλες ε, τέτοιου είδους εγκληματικές δραστηριότητες. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου τέτοιο χαρτόμισμα, αλλά να δώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπο. Σας ευχαριστώ για την πληροφορία που μου δίνετε, λέει η κυρία Επίτροπος. Θα το δούμε το θέμα ε, και ίσως πράγματι μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη ε, και τη διαδρομή αυτών των χαρτονομισμάτων. Ε, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω αυτή τη στιγμή, αλλά θα το δω το θέμα. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Υπήρξατε κατατοπιστική και κυρίως ειλικρινής στην απάντηση τη συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά την ημερομηνία ε, μέχρι μέχρι το σημείο που έχετε στοιχεία, δηλαδή μέχρι το 2007. Η ερώτηση αυτή ε, σας υπευλήθη από εμένα στις 6 Απριλίου του 2010. Στις 5 Μαΐου του 2010 στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, χάθηκαν άδικα, τραγικά, τρεις άνθρωποι κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων των Ελλήνων πολιτών που διεκδικούσαν ένα καλύτερο αύριο η ερώτηση ε, την επαναλαμβάνω για να αν μπορώ να έχω κάτι πιο συγκεκριμένο σχεδιάζει η επιτροπή να έχει ε, πιο ε, συστηματική παρέμβαση αν θέλετε και και συστάσεις στα κράτη μέλη για τα θέματα αυτά. σκοπεύετε πιο άμεσα και, και γρήγορα να συγκεντρώσετε στοιχεία για τα θέματα αυτά με δεδομένο ότι φαίνεται ότι το πρόβλημα εντείνεται ιδιαίτερα την περίοδο αυτή σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον εξώτομο κύριο Βουλευτή ότι βέβαια η Κομισιόν και εγώ προσωπικά πραγματικά εθλίβην ιδιαίτερα για το θάνατο των τριών αυτών ατόμων. Ήταν μια φοβερή τραγωδία όπου αθώοι χάθηκαν. Λυπούμεθα και οι σκέψεις μας με τις οικογένειες των θυμάτων αυτών. Όπως είπαμε θα πρέπει να εξετάζουμε και να συνεχώ συνεχώς τις στατιστικές μας. Η Eurostat το εξετάζει και ελπίζω θα μπορέσουμε μέσα σε αυτό να κάνουμε μια καλύτερη αξιολόγηση προσεχώς. Εμείς δεν σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή κάποιες πρωτοβουλίες από το θέμα, γιατί αυτή θα είναι διεμένη φρικτή, αλλά είναι πολύ περιορισμένη η αρμοδιότητα της Κομισιόν σε διαμεθοριακά εγκλήματα. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή σας λέω δεν προβλέπεται κάποια σχετική πρωτοβουλία. Thank you. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση υπαριθμών 22 του κ. Πότς όσον αφορά την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των θεωρήσεων διαβατηρία. Ε, Επίτροπος, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε, ξέρουμε κύριε Βουλευτά. Η πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναδομένη. Η κοινή πολιτική βασίζεται σε τρία νομικά ε, μέσα που εφαρμόζουν τα κράτη 531 του 2001 που αναφέρονται οι υπήκοοι των τρίτων χωρών που πρέπει να έχουν θεωρήσει και εκείνοι όχι. Δεύτερον, ο κώδικα θεωρήσεων διαμετριών που αναφέρονται όνοι οι όροι. Και τρίτον, ο κανονισμό 1683 95 που αναφέρεται στην μορφή, στην ενιαία μορφή των θεωρήσεων. Ο πρώτο οργανισμό στον οποίο αναφέρθηκα αναφέρεται σε ένα κατάλογο τρίτων χωρών που πρέπει να έχουν ε, θεώρηση διαβατηριών για να περάσουν σύνολα. Είναι ο συνεχόμενο αρνητικό κατάλογο και υπάρχει και ο θετικό κατάλογο των χωρών που εξαρτώνται βάσει κάποιων κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι και η αμοιβαιότητα. Αυτό ο οργανισμό αναφέρεται και να εφαρμόσουμε σε όλα τα κρατημένα εκτό από το Νόμο Βασίλειο και την Ελλαδία, καθώ επίση την Ισλανδία, την Νορβηγία και την Ελβετία. Βάσει αρχή αμοιβαιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι όσον αφορά του υπηκόου ε, από τρίτε χώρε που εξαιρούνται να ε, έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί όριο των διαβατηρίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι και οι υπήκοοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να απαιτούνται να έχουν ε, θεώρηση των διαβατηρίων του. Εάν υπάρχει εξέλιξη για κάποια κράτη-μέλη, ε, θα πρέπει παρόλα αυτά να επιβληθεί ο κανόνας της αμοιβότητας και ε, θα μπορούσε στην περίπτωση που δεν σημαίνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνει ή να προβλέψει μέτρα κατά των υπηκών των κρατών αυτών που απαιτούν παρόλα αυτά την θεώρηση. Βάσει του μηχανισμού της αμοιβαιότητας που εφαρμόζεται από το 2005 υπήρχαν 95 ε, περιπτώσεις ε, που αφορούσαν 13 χώρες του θετικού καταλόγου. Εν τω μεταξύ όμως υπάρχουν αμοιβαιότητα όπως η Ιαπωνία, Παναμά, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Ουρουγουάη και Κωνσταντίνα. Και πρόσφατα η Κομισιόν ολοκλήρωσε τις ε, διαπραγματεύσεις για την κατάργηση της ε, θεώρησης των διαβατηρίων με τη Βραζιλία και θα σας υποβληθεί αυτό σε εσά και στην, ε, στο Συμβούλιο. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα για κάποια κράτη-μέλη έναντι των ΗΠΑ και του Καναδά και είναι ένα θέμα που το συζητάμε αυτές τις ενόγω χώρες. Ο μηχανισμός αυτός δεν ισχύει στην περίπτωση των κρατών που βρίσκονται στον αρνητικό κατάλογο στην περίπτωση στην οποία το τρίτη χώρα αυτή εφαρμόζει διαφορετικού όρου για διαφορετικά κράτη-μέλη. Το κοινοτικό κεκτημένο δεν προβλέπει κανόνε για αυτέ τι περιπτώσει και ούτε προβλέπει ειδικού μηχανισμού και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Σπότ. Συμπληρωματική ερώτηση, 30 δευτερόλεπτα. Ναι, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που εγγυάται την ευρωπαϊκή πολιτική θεωρή στο διαβατήριο. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας και αν πραγματική αυτή η πολιτική βασίζεται σε αμοιβαιότητα θα ήθελα να ξέρω πόσο ακόμα θα δεχθεί η Κομισιόν την ε, ασύμετρη εφαρμογή των μέσων από τον Καναδά που υποβάλλει τους ε, Τσέχους την ανάγκη θεώρηση των διαβατηρίων. Επίτροπο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζω βέβαια την περίπτωση στην οποία αναφέρεται ο κ. Βουλευτή και η Κομισιόν έχει δεσμευτεί σε αυτό το θέμα. Οι Καναδικέ Αρχέ έχουν τώρα ε, μία υπηρεσία στην Πράγα. Ήταν αυτός ένας όρου που είχαμε πολύ και επίση έχουν και έναν οδικό χάρτη για την επαναφορά της ε, κατάργηση τη ε, θεώρηση των διαβατήριο είχαμε από κάποιε επαφέ υψηλού επίπεδου με το Καναδά, τι Τσεχικέ Αρχέ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Καναδοί είπαν να θα αλλάξουν το σχετικό νόμο και θα το υποβάλουν πολύ σύντομα στην Βουλή του. Βρισκόμαστε σε διάλογο μαζί του και με τι Τσεχικέ Αρχέ για να φροντίσουμε ο διάλογο αυτό να υπάρχει, ότι υπάρχει επικοδομητική ατμόσφαιρα και ότι μπορούμε πραγματικά να κινηθούμε προ μια επίλυση του προβλήματο και αυτό θα συζητηθεί εκ νέου στα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο στις αρχές Ιουνίου. Λυπούμε που δεν έχει επιληθεί ακόμα το πρόβλημα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι καταβάλουμε προσπάθειες για να βρούμε μια λύση το γρηγορότερο δυνατόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση, παριθμό 23 του κυρίου Χουντή για τις κοινέ δηλώσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας της 5ης Δεκάτου 2009. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Μάλιστα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά έχω σήμερα, ναι. Κύριε Βουλευτά, θα ήθελα πραγματικά να υπενθυμίσω ότι έχουμε δύσκολα παρελθόν διαπραγματεύσει με την Τουρκία που άρχισαν ήδη από την εντολή του 2002. Πρόσφατα όμως υπήρχαν πάρα πολλά θετικά βήματα που καταπληκτήκαν πέρσι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την παράνομη μεταρρύθμιση που έλεγε θα πρέπει να επιτευχθούν οι διαπραγματεύσει με την Τουρκία και πέρσι ο προκαταρχός Μίκος Μπαρό και ο Υπουργό Κατώνων Σουηδίας επισκέφθηκαν την Τουρκία και υπήρχε τότε μια δήλωση για πρόοδο. Υπήρξε εν τω μεταξύ πρόοδος, υπήρχαν διάφορες συνομιλίε. Από τότε και βρισκόμαστε τώρα πλησίων μία συμφωνίας για την ε, ε, ολοκλήρωση αυτών των συμφωνιών. Ε, προσπαθούμε να τελειοποιήσουμε αυτό το κείμενο το πλευρό των δυνατών και βέβαια έχουμε συνεχείς επαφές με τις ιστορικές αρχές. Ο στόχος μας είναι να τελειοποιήσουμε το θέμα και να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα διαπραγματεύσεων κατά διάρκεια της του Ιουνίου και θα κρατήσουμε βέβαια πλήρως ενημερό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια που έτσι θα πρέπει να εγκρίνει τα συμπεράσματα. Όσον αφορά τώρα το Frontex, δεν υπάρχει καμία αλληλένδεση μεταξύ αυτού και της ολοκλήρωσης ε, επαναφοράς της ε, ε της ε, Συμφωνίας Τουρκίας ΕΕ. Η Κομισιόν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σχολιάσει στην οριοθέτηση του επικράτειας ή των συνόμων ενό κράτους μέλους, μα αυτό είναι ε, θέμα του κράτους μέλους και βασίζεται στον διεθνή, στη διεθνή νομοθεσία. θα πρέπει να υπάρχει βέβαια μια συμφωνία προτού γίνει οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Ο κ. Χουντής έχει το λόγο. Τρία δευτερόλεπτα. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, από τη δυσκολία σε επανειλημμένες παρόμοιες ερωτήσεις να δώσετε πιο σαφή απάντηση, αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι διαπραγματεύσει σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολε. και κατά τον προσωπικό μου ισχυρισμό επιβεβαιώνει το ερώτημα ότι τίθενται πολιτικά ζητήματα από την πλευρά της τουρκίας που δυσκολεύουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. σας ευχαριστώ για την προθυμία σας που μόλι τελειώσουν αυτέ τι διαπραγματεύσει υπάρχει συμφωνία ευρωπαϊκή ένωση τουρκία θα είμαστε ενήμεροι. θα ήθελα λοιπόν συμπληρωματικά να σα πω το εξή πρόσφατα κατά την επίσκεψη του τούρκου πρωθυπουργού στην ελλάδα στην αθήνα υπεγράφει ένα πρωτόκολλο ένα μνημόνιο συνεργασία για θέματα παράνομη μετανάστευση με την ελλάδα. η ερώτηση που θέλω να σα κάνω είναι αυτό το μνημόνιο αυτή ας πούμε η συμφωνία επανεισδοχη μεταξύ και Τουρκία μπορεί να υποκαταστήσει την υποδιαπραγμάτευση συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης και τουρκίας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμπληρωματική ερώτηση. Δεν ξέρουμε τις ε, λεπτομέρειες ε, σχετικά με τη συμφωνία με μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Νομίζω όμως ότι αυτά αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε σε κάποια επικοδομητική διαδικασία. Υπάρχουν παράλληλα διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και όπως σας είπα είμαστε πολύ κοντά στο να το ολοκληρώσουμε το θέμα. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί είναι επικοδομητική και αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να το κλείσει το θέμα, αλλά και οι Τούρκοι μοιάζουν να θέλουν να συμφωνήσουν μαζί μας για την επανεισδοχή, γιατί κάτι τέτοιο θα είναι προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, ερώτηση. Κύριε Επίτροπε, και σε άλλες απαντήσεις που έχουμε λάβει, αναφέρεται ρητά ότι η Frontex διαπραγματεύεται με την Τουρκία τεχνικά ζητήματα. Αυτό το καταλαβαίνω. Ε, εσείς μας είπατε πρόσφατα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που ήσασταν μαζί μας και μας ενημερώσατε ε, για τα θέματα της αρμοδιότητός σας ότι η τελική συμφωνία με την τουρκία για τα θέματα παράνομη μετανάστευσης βρίσκεται όπως είπατε και σήμερα σε ένα πολύ καλό επίπεδο και φτάνει στο τέλος της. σε αυτή τη συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης και τουρκίας δεν πρέπει να υπάρχει πρόνοια και για τη frontex μεταξύ της ευρωπαϊκής ένωσης και της τουρκίας. δεν είναι η frontex ένας παράγων πολύ σημαντικός για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Ε, δεν ξέρω πόσα μπορείτε να μα πείτε από αυτά που περιλαμβάνονται στι διαπραγματεύσει όμω η κοινή λογική λέει αυτό δεν πρέπει εκεί να υπάρχει πρόνοια για την λειτουργία και τη δράση της Frontex. Ευχαριστώ πολύ. Yes, Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είχα τη δυνατότητα ε, την ε, περασμένη Δευτέρα να απευθυνθώ στην ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και ε, τότε είπα και επιμένω ότι έχει σημειωθεί πρόοδο στι διαπραγματεύσει με την Τουρκία. Όσον αφορά στη Frontex και στου ε, συνοριακού ελέγχου ε, τη Τουρκία, έχει επιτευχθεί μια αρχική συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Οι συζητήσει συνεχίζονται και προ το παρόν η Frontex περιμένει μια απάντηση από την Τουρκία για να συνεχιστούν οι συζητήσει. Βεβαίως η Frontex είναι σημαντικός παίκτη σε αυτό το θέμα, αλλά ε, κάθε πράγμα στον καιρό του. Πρώτα η συμφωνία και η παράλληλη συζητήση με τη Frontex, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο συζητήσεων. Επόμενη ερώτηση από την Βαρόνη Λάτφορτ ε, αφορά ε, στην... πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντιμοκρατική και τις παραδόσεις κρατουμένων της CIA. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Όπως ξέρετε το θέμα αυτό με ενδιαφέρει και έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν για το θέμα αυτό. Είναι σαφές ότι η ελευθερία και η ασφάλεια ε, συμβαδίζουν και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, βρίσκεται ε, στην, στον πυρήνα των προσπαθειών μας. Πάντα λοιπόν πρέπει να προσπαθούμε με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα. Και αυτό δεν είναι μόνο νομική προϋπόθεση αλλά και ένα βασικό στοιχείο για να προάγεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα αρχές και με τους πολίτες. Η ε, Κομισιόν λοιπόν ε, συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα, τη νομική αποτελεσματικότητα με τη σαφή δέσμαυση να γίνονται σεβαστά ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πρακτικές που αφορούν παραδείγματος χάρη στην παράνομη παράδοση κρατουμένων, αυτά είναι παραβίαση. Αυτό το έχει πει πάντα η Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη λοιπόν καλούνται να ε, διεξάγουν ανεξάρτητες έρευνες για να διαπιστωθεί η αλήθεια. Αυτή είναι μια υποχρέωση που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έτσι ώστε τα θύματα να μπορούν να αποκτήσουν αποζημίωση. Εμείς ε, έχουμε ενθαρρυνεί την Πολωνία και τη Ρουμανία να ε, κάνουν έρευνες σχετικά με τέτοιου είδου παράνομες παραδόσεις και επίση, ε, τον Μάρτιο του 2008 χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Πολωνία έλαβε τα απαραίτητα μέτρα. Η Λιθουανία και αυτή επιθυμεί να ξεκινήσουν έρευνες. Όσον αφορά τη συζήτηση για τις παράνομες αυτές πτήσεις και τις επιπτώσεις στην πολιτική αεροπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν ε, έλαβε το μαθημά στον τον Ιανουάριο του 2008 και επιπλέον ο ενιαίος ευρωπαϊκός ε, ουρανός ε, που τέθη πέρυσι επιτρέπει τον έλεγχο των αεροσκαφών και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό προσεκτικά. Το 2008 η Κομισιόν ε, προσέφερε πληροφορίες στο έγγραφο για την τρομοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτό αποτελά, αποτελεί ε, μια προσθήκη στον αγώνα κατά της ε, τρομοκρατίας. Όλα τα κράτη-μέλη απάντησαν σε αυτό το ερωτηματολόγιο και τώρα λοιπόν από πλευράς Κομισιόν ε, κάνουμε απολογισμό των βασικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρωτοβουλειών στον τομέα της αντιτρομοκρατίας μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Οι αντιτρομοκρατικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη αυτά δεν θα αξιολογηθούν ειδικά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σαφές το τι πιστεύει η Κομισιόν και εμεί θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων και των νομικών ε, προκλήσεων. Ε, θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε πολλά πράγματα ε, από βιώσιμες πολιτικές σε κοινοτικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι σαν να ψάχνουμε ψήλους τάχυρα. Σίγουρα θα πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε. Θα πρέπει η Κομισιόν να παρακολουθήσει το θέμα πιο στενά. Ωστόσο, στο παρελθόν κράτη-μέλη συμμετείχαν σε αυτή την παράδοση κρατουμένων. Άνθρωποι εξαφανίστηκαν και υπάρχει ένα τεράστιο κενό χάσμα μεταξύ των λόγων και της πραγματικότητας. Δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες, δεν έχει αποδοθεί λογαριασμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων δεν θα πρέπει να ασχολείται μόνο με την μελλοντική εξασφάλιση ε, των δεόντων, αλλά θα πρέπει να διερευνήσουμε και αυτά που έγιναν στο παρελθόν και αναφέρομαι και στην ε, κυβέρνηση του Νεμένου Βασιλείου μεταξύ άλλων. Τι θα κάνει η Επιτροπή για το παρελθόν. Κοίταξε, λέει η Επίτροπο, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δουλέψει πολύ επικοδομητικά, έχει δουλέψει πολύ σημαντικά και έχει ε, ρηχθεί φως αν θέλετε. Έχει χυθεί το φως σε αυτό το θέμα των παραδόσεων κρατουμένων και όντως η κοινή γνώμη θέλει να μαθευτεί η αλήθεια και εμείς ως Επιτροπή ενθαρρύνουμε πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των θεμάτων αυτών ε, στις χώρες και ε, το παρακολουθούμε και ζητούμε να γίνει. Έχουμε και την πρόταση για τον Ευρωπαϊκό Ουρανό και θα μας βοηθήσει να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά στο μέλλον. Θα το δούμε, θα ασκούμε πίεση για περισσότερη σαφήνεια, περισσότερη διαφάνεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά συγκεκριμένα πράγματα ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα συνεργαστούμε στενά ώστε να αποτελέσει αυτό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο κύριος Ζένεκερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα η κυρία Επίτροπος να μας πει κάτι το σημαντικό. Ε, έχουμε αυτή την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερωτώ λοιπόν κυρία Επίτροπε, θεωρείτε ότι τα κράτη-μέλη τίνουν περισσότερο στην συνεργασία μοιράζονται όλο και περισσότερο στοιχεία λεπτά, πληροφορίες ε, ε, τέτοιου είδους για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Κάνουν βήματα προς τα εμπρός προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια είναι η άποψή σας κυρία Επίτροπε. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όντως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι κάτι το πολύ σημαντικό ε, και βεβαίως τις σημαντικές δράσεις τις ε, υλοποιούν οι εθνικές αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις πρωτοβουλίες αυτές, προσφέρει ένα νομοθετικό πλαίσιο, ε, ε, ασκεί πίεση έτσι ώστε να τηρηθεί η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχουμε χρηματοδότηση, μπορούμε να προσφέρουμε στήριξη στα θύματα και μπορούμε να ενθαρρύνουμε περαιτέρω συνεργασία. Έχω την αίσθηση ότι πολλά γίνονται ε, στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Βεβαίως ε, υπάρχει το πολύ λεπτό ζήτημα του μοιράσματο ε, προσωπικών και λεπτών των και απόρριτων, αν θέλετε, πληροφοριών είναι ένα ζήτημα που εξαρτάται απόλυτα από την ύπαρξη ή μη αμοιβαία εμπιστοσύνη από τη διασφάλιση ότι όλα τα ε, ένομα συστήματα ε, σέβονται το κράτος δικαίου και αξίζει να τα εμπιστευτεί ο ΜΕΝ τα συστήματα που έχει ο ΔΕ. Σίγουρα έχει έχουν εκφράσει τη βούλησή τους στα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θέλουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, σεβόμενοι πλήρως όμως ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο για τις ε, πολύ ε, ακριβείς και συγκεκριμένες απαντήσεις που έδωσε ε, σε, ένα, σε, πολύ, σε πολύ δύσκολα και περίπλοκα θέματα. Έχουμε τώρα τις ερωτήσεις υπαριθμών 25, 26 και 27. Ε, κυρία Μακίνες, συγγνώμη Πρόεδρε που σας διακόπτω. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε ποιες ερωτήσεις θα απαντηθούν η ερώτηση 33 ας πούμε θα απαντηθεί γιατί όλοι πρέπει να πάμε και σε άλλες συνεδριάσεις. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιες ερωτήσεις δεν θα απαντήσετε. Ο πρόεδρος, είναι εξαιρετικά πιθανό να φτάσουμε στο ερώτημα υπαριθμό 33. Αν περιμένετε γι' αυτό ίσως δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε τώρα 8 ερωτήσεις, δεν πρέπει να προλάβουμε και δεν θα φτάσουμε στην 33. Έχουμε λοιπόν 8 ή 7 διορθώνω λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε ερωτήσεις και ο κύριος Σταγιάννη θα απαντήσει από κοινού, θα απαντήσει για όλες αυτές τις ερωτήσεις μαζί. Έχετε το λόγο. Να σας πω καταρχάς ότι θα τελειώσουμε στις 8 και γιατί ε, θα πρέπει και οι διερμηνείς ε, να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα ε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στις 9 το βράδυ στη συνέχεια. Κύριε Ταγιάννη, έχετε το λόγο λοιπόν να απαντήσετε για όλες τις ερωτήσεις που σας έχουν απευθυνθεί από μαζί. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πάντοτε ε, μου ασκείτε πίεση να είμαι σύντομος, έχω πλέον συνηθίσει. Έχουμε λοιπόν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διάφορες ερετήσεις για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε και το καθήκον να ε, προλάβουμε έτσι ώστε η οικονομική κρίση να μην μετατραπεί σε κοινωνική κρίση και να μην πληγούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλοι όσοι εξαρτώνται από αυτούς. Από αυτές. Έχουμε την πρωτοβουλία λοιπόν για τις μικρές επιχειρήσεις, Small Business Act, και έχουμε νομοθετικές ε, προτάσεις που θα υπάρξουν Έχουμε κανονισμό για τις ε, κρατικές ενισχύσεις, για τις κυρώσεις, για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, για τις έγκαιρες πληρωμές. Όλα αυτά τα αιτήματα υπάρχουν και για το ενιαίο καταστατικό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ε, πέρα από αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουμε και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες. Έχουμε κάνει διάφορες μελέτες σε αξιολόγησης επιπτώσεων και πάντοτε εξετάζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Τα κράτη-μέλη εκτός αυτού έχουν δείξει ότι έχουν ισχυρή πολιτική βούληση ε, για να εφαρμοστεί αυτή η, ε, αυτός ο νόμος περί μικρών επιχειρήσεων. Παραδείγματο χάρη έχουν συμπεριλάβει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στις εθνικές τους αποφάσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν ανάμεσα στους βασικούς αποδέκτες των μέτρων που έλαβαν τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Παραδείγματο χάρη, η δημιουργία των ε, συστημάτων ε, για την χορήγηση δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά είναι από τα μέτρα που ελήφθησαν για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Εξάλλου, ε, η μέθοδοι αυτή ε, δείχνουν ότι είναι σωστός ο δρόμος, γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το νόμο περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και επίσης οι πράξεις που συστήνονται να υλοποιηθούν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η πολιτική προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, έχει άμεση σχέση και με τη στρατηγική περί Ευρώπης 2020. Αποτελεί άμεσο ε, στοιχείο αυτής και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί και αυτή στη στρατηγική των κρατών μελών. Μία από τις οδηγίες που έχουν ε, προταθεί από την κρατημέλη έχουν ακριβώς ως στόχο να βοηθηθούν τα κρατημέλη να υιοθετήσουν μία σειρά μέτρων προ όφελο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με βάση τις αρχές του Small Business Act επόμενη φάση θα είναι εκείνη όπου τα κράτη-μέλη θα κληθούν να υιοθετήσουν τα μέτρα αυτά στα εθνικά τους προγράμματα. Κατά το τέλος αυτού του έτους ε, κατόπιν θα υπάρξει ενδελεχής έλεγχος ε, της εφαρμογής του νόμου για να μετρηθεί η πρόοδος που θα έχει επιτευχθεί και για να ληφθούν νέα μέτρα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους τις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020. Ανάμεσα στις δράσεις που θα προταθούν θα είναι βελτίωση στην πρόσβαση για την πίστη και για την ανανέωση, δράσεις για ανανέωση του επιχειρηματικού πνεύματος και προαγωγή της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, κυρίως εκείνες ε, ε, τις οποίες διαχειρίζονται νέοι επιχειρηματίες είναι οι βασικοί αποδέκτες αυτών των νέων πρωτοβουλειών. Γνωρίζοντας πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή για να αποκτήσουν δάνεια, ε, αυτό το ξέρει αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να εφαρμοστούν έλεγχοι και έρευνες για την κατάσταση. Και η Κομισιόν έχει επεξεργαστεί και μία σειρά προγραμμάτων που προσφέρουν οικονομική ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αποκτήσουν και αυτές πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τι δραστηριότητέ του. Το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, παραδείγματο χάρη, συγκεντρώνει διάφορα οικονομικά εργαλεία τα οποία διατίθενται μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για εγγύησει ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα Ζερεμής προσφέρει ένα μεγάλο γκάμα οικονομικών εργαλείων συγκεκριμένων έτσι ώστε να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην ε, ευρωπαϊκή επικράτεια. Και τέλος το νέο αυτό εργαλείο των μικροπιστώσεων αυτή είναι μια ιδέα κοινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τράπεζας Επενδύσεων έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν δυσκολίες να αποκτήσουν δάνεια. Η πρόσβαση των μικρομεσαίων στην ε, πίστη αυτή ε, έγινε δυνατή λόγω της γραμμής προεπολογισμού που συμφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις ενδιάμεσες τράπεζες στις οποίες είχε ανατεθεί και αυτές να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μορφή δανείων. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφώνησε σε 13 δις ευρώ ενίσχυση. Αυτό λοιπόν ισοδυναμεί με αύξηση 55% σε σχέση με την ε, προηγούμενη χρονιά πάνω από 70% των 21 ε, ε, δισεκατομμυρίων που συμφωνήθηκαν για το χρονικό διάστημα 9 μέχρι 11 αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή 50 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η Επιτροπή πριν από κάποιες ημέρες, ε, πρόσφατα δηλαδή, οργάνωσε μια συνεδρίαση, ένα συνέδριο που ε, συναντήθηκαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα συνέδριο όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί συμφωνήθηκε να εξεταστεί η κατάσταση στην αγορά και να ζητηθούν νέες στρατηγικές έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση. Έπρεπε λοιπόν να, στηθεί, ε, να στηθούν μέτρα έτσι ώστε να βελτιωθεί η οικονομική ανάκαμψη. Και μία από τις αποφάσεις που λήφθησαν είναι να υπάρχει ένα μόνιμο φόρουμ συζητήσεων όπου θα είναι παρόντες οι οικονομικοί οργανισμοί, ε, τα ταμεία ε, κεφαλαίου κινδύνου προβλέπονται και με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τριμηνιαίοι έλεγχοι. Ε, στο φόρουμ αυτό θα διαπιστωθεί η πρώτη φάση μιας στρατηγικής που θα έχει ως στόχο το πώς ακριβώς προχωράει η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων οχήσεων στην ε, Ένωσή μας. Και τέλος, ε, δράτω με αυτή τη ευκαιρία για να σας ενημερώσω ότι στο πλαίσιο της ε, πρώτης εβδομάδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα λάβουν χώρα πάνω από 1.200 εθνικές εκδηλώσεις και σε περιφερειακό επίπεδο για πολλά θέματα που αφορούν ε, αυτόν τον τομέα. Την ε, εβδομάδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή θα είναι 25 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, παράλληλα με την παράδοση ε, των ε, βραβείων των επιχειρηματικών που προβλέπεται αυτή στις 31 Μαΐου στη Μαδρίτη. Και όλα αυτά για να σας δείξω ότι εγώ προσωπικά στρατεύομαι έτσι ώστε η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση ε, λόγω της υποστήριξης που θα τύχουν οι μικροπεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να στηριχθεί γιατί είναι βεβαίως απαραίτητο να αναδιερθρωθεί η μεγάλη βιομηχανία. Αυτή θα οδήγησει στην απώλεια θέσεων εργασίας και ως εκ τούτου εμείς μπορούμε την απασχόληση να την επαναφέρουμε μόνο εφόσον ενισχύσουμε την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ράχο ράχο κοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να αλλάξω κάπου γιατί η Κομισιόν αν... ανέπτυξε την ερώτηση, την απάντησή της τόσο πολύ. Λοιπόν, μισού λεπτού συμπληρωματικέ ερωτήσει. Κυρία Χάρκιν, πρώτα. Ναι, σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Παρ' όλα αυτά, κύριε Επίτροπο, αναφέρθηκε ότι το πιο κέριο πρόβλημα είναι η πρόοδο στο κεφάλαια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έδωσε στην Ιρλανδία κάποια χρήματα, αλλά πολλά χρήματα δεν έχουν διανεμηθεί γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ των ανάγκων των ΜΜΕ αναχρηματοδότηση και των στόχων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που είναι επενδύσεις μέσω και βραχυπρόθεσμες. Τι θα γίνει λοιπόν με εκείνες τις ΜΜΕ που είχαν προηγουμένως χρηματοδότηση κατά αυτόν τον τρόπο και επίσης θα μπορούσατε να δώσετε κάποιε εγγυήσει όπω αυτό που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ λοιπόν, κύριο Σίγκεντ. Σίγκεντς. Θα ήθελα να σα πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριο Επιτροπό ότι οι ΜΜΕ είναι πάρα πολύ σημαντικέ <clears throat> στην οικονομία και όχι μόνο λόγω των θέσεων αποσχόληση που δημιουργούν αλλά και επίση γιατί ε, ε, είναι πιο σταθερέ. Ε, από ότι μεγάλες ε, επιχειρήσεις ε, που έρχονται ξαφνικά και δεν αφορούν σε κανένα. Συμφωνώ όμως με αυτά που είπε η κυρία Χάρκιν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Το ανέφερε και ο Επίτροπο. εκτό αυτού υπάρχει υπερβολικά πολύ γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Μίτσελ, Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω τον Επίτροπο κατά πόσον θα εξετάσει προβλήματα μη άμεση χρηματοδότηση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μην ξέρω τι στη χώρα σα. Στη δικιά μου χώρα δεν υπάρχει πια ένα μάνατζερ στην τράπεζα. Βλέπουν τα, τα χρήματα από τις τράπεζες δίνονται χωρίς καμία διαχείριση, χωρίς κανέναν έλεγχο. Δίνονται αυτόματα. Και αυτά είναι τα προβλήματα που είχαμε. Σε αν είχαμε μία συμπληρωματική θέση απασχόληση σε κάθε μία μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη, θα είχαμε λήξει το πρόβλημα της απασχόλησης. Σας παρακαλώ, για σκεφτείτε το και προσπαθείτε να μας αναφέρετε στους παραδοσιακούς μάνατζερ των τραπεζιών που έπαιζαν ένα ρόλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ευχαριστώ, κύριε Σέλβατ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Προφανή ερώτημα κατά πόσο η Κομισιόν πιστεύει ότι η εβδομάδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Μπορώ να ρωτήσω λοιπόν την Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνουν ώστε να είναι σίγουρο ότι ε, ανά την Ευρώπη οι επιχειρηματίε και οι οικογενειακέ επιχειρήσει θα επιζήσουν και δεν θα παρεμβολήσουμε τι μικρομεσαίε υπηρεσίε, αλλά θα τι ενδυναμώσουμε και τι ενθαρρύνουμε. Ευχαριστώ ο Επίτροπος μπορεί να απαντήσει πάρα πάρα πολύ σύντομα για να τελειώσουμε πραγματικά στη και Λοιπόν, έχετε πολλές ερωτήσεις, αλλά... Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία είπαν οι αξιότιμοι βουλευτές όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ε, συναντήθηκα με τον πρόεδρο Μάιστατ και τον κάλεσα ε, τα, τα 30 δις που είχαν προβλεφθεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή δυνατόν να τα διαθέσει το συντομότερο δυνατόν. Αυτή ήταν μια παρέμβαση που είχα προαναγγείλει και εδώ στο Κοινοβούλιο το οποίο βεβαίως ε, τότε μου προσέφερε την υποστήριξή του. Η απάντηση του Προέδρου ήταν ε, θετική και μου είπε ότι μετά από, ε, μια, από κάποιες αρχικές δυσκολίες έφτασαν 7 από τα 30 που προβλέπονται. Βεβαίω ε, θέλω να τον ξανακαλέσω να επιταχύνει λιγάκι την όλη διαδικασία έτσι ώστε το πρόβλημα που αφορά στις ε, τράπεζες όπως είπε και ο τελευταίος ομιλητής κατά κάποιον τρόπο να λυθεί. Γιατί το τραπεζικό σύστημα είναι διαφοροποιημένο. Δεν είναι ίδιε όλε οι τράπεζε. Υπάρχουν εκείνε που ασχολούνται με την κερδοσκοπία, αλλά ευτυχώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα δίκτυο τραπεζών όπου ο διευθυντή γνωρίζει τον επιχειρηματία που ζητάει δάνειο ε, και είναι και επίση σίγουρο ότι θα πάρει πίσω τα λεφτά του, έτσι ώστε να μην συμβεί αυτό που συνέβη στι ΗΠΑ το συνέδριο αυτό που όπως σας είπα οργανώθηκε πριν από λίγες μόνο ημέρες ε, και με τη συμμετοχή των δικών σας των συναδέλφων είχε ως στόχο να μελετηθεί μία ε, στρατηγική. Εμείς ε, συστήσαμε ένα φόρουμ για να χορηγηθούν πιστώσεις και Παραδείγματο χάνει για να είναι ανταγωνιστικέ οι επιχειρήσει πρέπει να είναι καινοτόμο. Όμω ε, καινοτομία δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρχουν και χρήματα. Ω εκ τούτου εγώ ε, θεωρώ ότι είναι πρώτο μου και πρωταρχικό μέλημα να συμπεριλάβω και τι τράπεζε στα προγράμματά μου. Και οι τράπεζε έχουν δεσμευτεί για το μέλλον. Ω εκ τούτου με ουσιαστική δράση και με κίνητρα πλευρά τη Επιτροπής όπου θα συμμετέχουν οι ε, τράπεζες, ε, οι επιχειρηματίε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία συμμετείχε με δυο τρει αντιπροέδρους στη συζήτηση. Με όλα αυτά έχουμε ως στόχο να ε, μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τουλάχιστον κάποιους στόχους γιατί σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι το καλύτερο εργαλείο για να βγούμε από την κρίση και όπω σα είπα για να αποφύγουμε η οικονομική κρίση να μετατραπεί και σε κοινωνική. Μπορείτε να βασίζεστε στην απόλυτη στράτευσή μου, έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προστατευθούν με την ελπίδα ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορέσουν να αναγεννηθούν γιατί στην ε, οικονομία της αγοράς αυτό που έχει σημασία είναι οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματική κοινωνική πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη τους συνέδρους που ήταν τόσο σύντομος ο χρόνος εργασίας αλλά είχαμε μια υπέρβαση στις προηγούμενες συνέδρε. μέσα στις 25 οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου θα απαντηθούν από τα τέλος της ερωτήσεων διακόπτη συνεδρίες με 9.